El señor Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κυρίζω την έναρξη της ε, Συνόδου για σήμερα Πέμπτη. Μετά από το χθεσινό αγώνα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται την έκθεση του κυρίου George Lyon σχετικά με το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής μετά το 2013. Και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ο Επίτροπος βρίσκεται ανάμεσά μας διότι γνωρίζω πως ε, αυτή την ε, εβδομάδα ε, Συναντήσαμε πολλούς επιτρόπους, αλλά δεν ήταν πάντα οι αρμόδιοι επί των θεμάτων που εξετάζαμε. Και μπέστο στην περίπτωση αυτή έχουμε τον αρμόδιο επίτροπο και αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο πρωτίστως στον κύριο George Lyon, ο οποίος ως συγητής αυτής της σημαντικής έκθεσης θα μας μιλήσει για τέσσερα λεπτά προκειμένου να παρουσιάσει την έκθεσή του και δύο λεπτά για να απαντήσετε στο τέλος της συζήτησης. Ο εισηγητής φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα έξι λεπτά στην αρχή του παρουσίαση, αλλά τότε θα του επομένει χρόνος προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις συναδέλφων και στους σχολιασμούς. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να χρησιμοποιήσει τα τέσσερα λεπτά αρχικά. Εν είναι κυρίω του εαυτού του και θα κάνει όπως νομίζει. Κύριε Λάιου, να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, ε, προσφέροντας τα συλληπιτήριά μου και τα συγχαρη... στους Γερμανούς συναδέλφους και τα συγχαρητήρια στους Ισπανούς συναδέλφους μετά από τον εξαιρετικό αγώνα. Θέλω να ξεκινήσω με τα δύο βασικά θέματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε από πλευράς της αναθεωρήσεως της ε, κοινοτικής γεωργικής πολιτικής. Τι αντιπροσωπεύει και ε, ποιε είναι οι προκλησει του 21ου αιώνα. Ε, υπάρχουν ε, προπολογισμοί λιτότητο και πρέπει να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη στήριξη των γεωργών και στο μέλλον. Ένα βασικό, μια βασική πρόκληση την οποία να αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι πώς θα αντιμετωπίσει την αύξηση της σε τροφίμων που σύμφωνα με τον ΠΟΕ θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050 έχοντας λιγότερη γη, ε, λιγότερο νερό και λιγότερη ενέργεια λόγω ε, των κλιματολογικών αλλαγών. Και ε, ο Sir John Μπέντιγκτον είχε πει το 2009 σχετικά με τις θεομηνίες ότι θα έχουμε μία θεομηνία τεράστια το 2030 και αν δεν αντιμετωπίσουμε τα θέματα που τίθενται τότε θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα ιδίως ε, μετανάστευσης διότι πολλοί θα μετακινηθούν για να αποφύγουν τις ελλείψεις ύδατος. Πρέπει λοιπόν έτσι να έχουμε μία πιο βιώσιμη γεωργία και η στόχη αυτή πρέπει να είναι στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης για να μπορέσουμε μπορέσουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους Ευρωπαίους πολίτες μας και να ναι. και να ε, ε, συνεχίσουμε να ε, παράγουμε και τα βιολογικά καύσιμα και τα τρόφιμα για να στηριχθούν οι, οι γεωργοί. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει προστασία για να μπορέσουν οι γεωργοί να συμμετάσχουν στα προγράμματα και οι γεωργικές εκτάσεις να καλυφθούν από αυτά τα προγράμματα στην επόμενη αναθεώρηση. Και τέλος πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, τους γεωργούς ε, και ε, περισσότερο από ό,τι να τους τιμωρούμε και να τους απειλούμε. Ιδίω στα νέα κράτη θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή στις άμεσες πληρωμές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα πρέπει να σταματήσουν οι ε, πληρωμές το 2020 ε, σε σχέση με το σχήμα που υπήρχε προ 10 ετών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει μια δικαιοσύνη και ισότητα που να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Θα αντιμετωπίσουμε και την αστάθεια των αγορών. Χρειαζόμαστε πρόληψη και αποθήκη πρέπει να ασφαλίζουμε και να ε, μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις μελλοντικέ αγορές αλλά δεν πρέπει να επανέλθουμε στις παλές μεθόδους του παρελθόντος διότι θα ήταν σωστό να μην επανέλθουμε σε αυτό το παρελθόν. Είμαι αισιοδόξος ότι το Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει τους στόχους μας, να εξυγχρονίσει την κοινή γεωργική πολιτική, να την προσαρμόσει στους στόχους του 21ου αιώνα και ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συζητήσει και να διαγράψει ένα πρόγραμμα δράσεως και ε, καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αναθεωρήσει τις προτάσεις της όταν θα τις δημοσιεύσει τον Νοέμβριο. Ευχαριστώ κύριε Λάιν. Ο κύριος ε, Επίτροπος Χιόλος έχει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ε, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που συμμετέχω σε αυτήν τη συζήτηση, διότι θα πρέπει να κάνω προτάσεις για τη μετέθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και όπως το είπα για κατά τη διαρκεία των ακρόασεων στο Κοινοβούλιο, οι σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι είναι θεμελιώδες προκειμένου να καταλήξουμε στο τέλος σε μια μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θα ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες των πολιτών και θα γίνει ακόμη καλύτερα κατανοητή από τους πολίτες της Ένωσης. Ευχαριστήσω τον George Lyon για την έκθεση που συνένταξε και μας υποβάλλει σήμερα, φυσικά με όλο το επιτελείο του, όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, αγροτικής πολιτικής μέσω τροπολογιών των οποίων ε, μπλουτίστηκε το κείμενο. Ε, τονίζω επίσης ε, την ε, ανάγκη μιας καλύτερης επικοινωνίας πάνω σε τα αγροτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι πέραν κάθε τεχνικής φύσης λεπτομέρειας της εκθέσης, η έκθεση αυτή είναι να πολύ καλό μέσο για να επικοινωνήσουμε επί θεμάτων αγροτικής πολιτικής, διότι η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να ε, προβλέπει και να προλαμβάνει τις εξελίξεις του μέλλοντος. Επίσης ε, θα ήθελα να σας ε, ζητήσω πως θα πρέπει να ευθερμαστούμε όχι μόνο με την συνθήκη της Λισαβόνας που βλέπει τις μου στόχους για την ΚΑΠ αλλά και για τη συνθήκη της Ευρώπης σχετικά με το 2020. Ε, έχουμε την ευκαιρία εδώ προκειμένου να προσαρμόσουμε καλύτερα την κοινή αγροτική μας πολιτική στις προσδοκίες των πολιτών πέραν αυτών των παραδοσιακών στόχων το να διασφαλίσουμε την ε, ε επιστηστική ασφάλεια και τροφοδοσία των αγορών. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και την ε, τροφική αλυσίδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών, την διαφάνεια την οποία απαιτούν η ε, παραγωγή και οι καταναλωτές. Αυτό βρίσκεται μόνο στο πλαίσιο της μερινή ΚΑΠ, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει και θα προτείνει η Επιτροπή. Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την εκθεσή σχετικά με τις άμεσες ε, ενισχύσεις, ε, κάτι το οποίο μπορεί να διασφαλίσει όχι μόνο τη σταθερότητα των εισοδημάτων των γεωργών, αλλά να διασφαλίσει επίσης και ένα ελάχιστο επίπεδο για την ε, ε, σε επίπεδο σε ζητήματα δημόσιων αγαθών. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ένα ελάχιστο εισόδημα των γεωργών αλλά και να τους παροτρύνουμε προκειμένου να ε, παράγουν δημόσια αγαθά. Επίσης ε, είδα την πρόταση σας σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος ε, άμεσων ενισχύσεων για να διασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ισότητα ανάμεσα στις κατανομές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και στις κατηγορίες των γεωργών λαμβάνοντας υπόψη την, ε, ε την ιδιαιτερότητα των γεωργών που ζουν και εργάζονται σε περιοχές ε, ορεινές ή προβληματικές. Επίσης χρειάζεται να υπάρξει μια, ένας προσανατολισμός ο οποίος θα οδηγήσει σε μια βελτίωση των ε, αγορών στι οποίες απευθύνονται οι γεωργοί. Θεωρώ πως η βελτίωση των μηχανισμών διαχείρισης των αγορών είναι κάτι το κατάλληλο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι αγορές και να μην επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων που έχουμε, δηλαδή να διατηρήσουμε την γεωργία σε όλη την ε, νοσιακή επικράτεια και να βοηθηθούν έτσι οι γεωργοί μας. Και τώρα μερικά σχόλια επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν και που πρόκειται να συζητηθούν. Ορισμένα σχόλια λοιπόν περί αυτών. Θεωρώ πως ε, παραγωγή τροφίμων είναι ένα σημαντικός στόχος της ε, ΚΑΠ που, η οποία αμείβεται κιόλας από την αγορά αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα δημόσια αγαθά που δεν ε, αμείβονται από την αγορά αλλά θα πρέπει να καλυφθούν από μια συμβολή του δημοσίου. Αυτέ οι δύο πτυχέ λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, την παραγωγή τροφίμων και την παραγωγή δημοσίων αγαθών με πτυχέ που αμείβονται από την αγορά και άλλες πτυχέ που υποστηρίζονται από, τον, από το δημόσιο, τον δημοσιοπροπολογισμό. Η δομή σε ό,τι φορά την κοινή πολιτική και επανειλημμένα το έχω τονίσει, έχει ανάγκη από δύο πυλώνε για να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, αλλά και μια διαχείριση πιο αποτελεσματική των μέσων που έχουμε στην διάθεσή μας, διότι έχουμε εργαλεία τα οποία εφαρμόζονται και, αξιο... και αξιολογούνται αλλά υπάρχουν και κάποια εργαλεία τα οποία έχουν πιο μακροπρόθεσμη διάρκεια και ως εκ τούτου ε, χρειάζομαστε περισσότερα χρόνια για να διασφαλίσουμε αυτήν την καλύτερη διαχείριση των πόρων ε, και των μέσων που έχουμε στην κοινή πολιτική. Οι δύο αυτοί πυλώνες λοιπόν είναι απαραίτητοι. Υπάρχει συμπληρωματικότητα λοιπόν των δύο αυτών πυλώνων αλλά και ένας σαφέστερος προσδιορισμός των στόχων τους και ο τρόπος εφαρμογής των εν μέτρων. Τώρα σε ό,τι φορά την ε, πολλαπλή συμμόρφωση, νομίζω ότι αυτό είχε θετικότερες επιπτώσεις ε, αναφορικά με τις άμεσες ε, επιδοτήσεις, τα μεσενισχύσεις, συγγνώμη. Φυσικά μπορούμε να απλουστεύσουμε τα μέτρα της πολλαπλής συμμόρφωσης, μπορούμε το περιεχόμενό τους να καταστεί σαφέστερο τόσο για τους ε, γεωργούς όσο και για τις ε, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις ε, που ελέγχουν, αλλά η πολλαπλή συμμόρφωση η οποία συνδέεται και με τις ενισχύσεις είναι ένας ε, σωστός τρόπος για να εκτιμήσουμε και το θέμα των ε, απόδοσης των δημόσιων αγαθών. Τώρα για τα μέτρα που λαμβάνουμε στις, ε, σχετικά με τις αγορές έχουμε ανάγκη από το να διατηρήσουμε και ένα δίκτυο ασφαλείας και να μελετήσουμε νέα μέτρα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στην επιτεύξη μιας σταθερότητας των τιμών και των εισοδημάτων στον κλάδο τώρα για τις ε, δομές μικρές, μεσαίες, μεγάλες εκμεταλλεύσεις και για τις, ακόμα και μικρές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να ε, βελτιωθούν και να τίνουν προς την ε, μεγαλύτερη αποδοτικότητα άρα μπορεί να υπάρξει αναδιάρθρωση αυτών των μικρών εκμεταλλεύσεων που θα συμβαδίσει με τις εξελίξεις των αγορών χωρίς ε, να μεταβούμε σε ένα ενιαίο μόνο γεωργικό μοντέλο. Να διατηρήσουμε λοιπόν την διαφορετικότητα, την πυκλομορφία που υπάρχει. Αυτά είχα να σας πω πλευρά μου. Περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας. Και κύριε Λάιον, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, θα ε, είστε βέβαιοι ότι θα κοιτάξω ε, αναλυτικά όλες τις ε, τροπολογίες ε, τις οποίες θα λάβει υπόψη σε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα λάβει η Κομισιόν τους προσεχείς μήνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Για ένα λεπτό το λόγο θα λάβει ο συνάδελφος Λαβία ως εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι αυτή η έκθεση Lion έχει το πλονέκτημα να έχει καθορίσει με σαφήνεια ένα σύνολο στόχων της κοινή αγροτικής πολιτικής ε, με στόχους πιο ευρύς από το παρελθόν σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσης για το 2020. Αυτή η γεωργική πολιτική φαίνεται διαφαίνεται από την έκθεση και θα πρέπει να παραμείνει η ρύθμισή της σε κοινοτικό επίπεδο. Θα τεθεί λοιπόν τροχοπέδι σε όλους εκείνους που προέβλεπαν μια επανεθνικοποίηση, εθνική υποστήριξη στην ε, αγροτική πολιτική. Ξαναφαίνεται ότι ζητούνται οι αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των στόχων, που είναι ευρύτεροι. Και χρειάζονται περισσότεροι πόροι και για την πρόθεση των δημοσίων αγαθών. Και φαίνεται από την έκθεση επίσης ότι οι πόροι που προορίζονται για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να ταιριάζουν ε, και με τα όσα είχαν τους στόχους που υπήρχαν κατά το παρελθόν για την κοινή αγροτική πολιτική. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχουν οι ομιλητές του των ομάδων του Κοινοβουλίου. Και πρώτα ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον George Lyons καθώς και την ομάδα των σχεδόν εισηγητών που εργάστηκαν νομίζω ε, με μεγάλη σύνεση συνέταξε την έκθεση και τίθενται φιλοδοξίες για την ε, ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Μετά την κρίση του 2007 και 2008 των πρώτων υλών και μετά την αγροτική κρίση του 2009 μάθαμε ότι ο φιλελευθερισμός δεν είναι η λύση για τη Γεωργία. Η Γεωργία έχει στόχο πρωταρχικό να προσφέρει, να εγγυάται μάλλον την επισητιστική βοήθεια για 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους αλλά θα πρέπει να έχουμε και εμείς και σε, τη θέση μας σε μια φερέγγια αγορά. Οι συνθήκες που επεκράτησαν από τα μέσα του 20ου αιώνα άλλαξαν. Οι τεχνικές άλλαξαν και θα πρέπει να αλλάξουν ακόμα. Και τα πολιτικά εργαλεία για την εργοτική πολιτική θα πρέπει να εξελιχθούν δεόντως. Η Γεωργία θα πρέπει να συνοδεύεται στην εξέλιξη αυτή. Αν ο πρώτος πυλώνας σηματοδοτείται μόνο από τον ευρωπαϊκό πυλώνα και πρέπει να καλύψει εξωτερικού στόχους, ο δεύτερος που συγχρηματοδοτείται θα πρέπει να συνοδεύει τον εξυγχρονισμό της γεωργία και του αγροεπιστημιστικού τομέα για να ληφθούν υπόψη νέε συνθήκε. Αυτή η πολιτική θα πρέπει επίσης να είναι δικαιότερη. Δικαιότερη λέω. Μεταξύ χωρών και μεταξύ των γεωργών. Εμείς τι θέλουμε, να ξαναδώσουμε ελπίδα στα 14 εκατομμύρια γεωργών και στις οικογένειές τους για να αντικαταστούν τα 4,5 εκατομμύρια γεωργών που είναι πάνω από 60 ετών σήμερα και που θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Το θέμα της ανανέωσης των γενιών και του πληθυσμού θα είναι μία από τις ε, προτεραιότητές μας. Εξ των σοσιαλιστών τον λόγο έχει ο κύριος Ολέσνιτζακ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε ε, ε, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση την οποία διεξήγαμε τους τελευταίους μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι χρειάζονται αλλαγές στην κοινή γεωργική πολιτική. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτή η κοινή πολιτική ε, θα πρέπει να εγγυηθεί στις επόμενες δεκαετίες την εξασφάλιση επαρκών τροφίμων αλλά να καλύψει και την βιοπικιλότητα και την διατήρηση της φύσεως. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε εις ε, τις ε, κοινωνικές επιταγές και να δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Ήπεθρο και η γεωργία θα πρέπει να έχει επαρκής, ε, ε, επαρκή έσοδα για να μπορέσει να ε, ανταμείψει την εργασία και να παραδώσει τα αγαθά και τα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη διάφορα θέματα. Έχουμε προκλήσεις για το μέλλον σχετικά με τις δαπάνες και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και των προμηθευτών και των παραγωγών και των καταναλωτών. Ευχαριστώ τον κύριο Λάιον για την έκθεσή τους. Για ένα λεπτό εξ των Σωμάς Φιλευθέρων, κύριε Πόλσαν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ο κύριος Λάιον κατόρθωσε να συντάξει μια έκθεση όπου αναφέρονται περικά σύντομα βήματα προς το μέλλον. Μικρά βήματα μεν, εξαιρετικά σημαντικά δε. Διότι αναφερόμαστε στην αλλαγή της αγροτικής μας πολιτικής. Χρειαζόμαστε βεβαίω μια κοινή αγροτική πολιτική, την χρειαζόμαστε και γι' αυτό δεν θα πρέπει να μιλάμε για επανεθνικοποίηση αυτής. Αυτό θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Να αφήσουμε εκτό αυτή την επιλογή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή, νέα εποχή, με πολλά δύσκολα, καθόδη θέματα που πρέπει να εξετάσουμε και είναι η υποχρέωσή μα να λύσουμε τα προβλήματα και τα θέματα αυτά. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπου, που πρέπει, ε, δισεκατομμύρια ανθρώπους που πρέπει να τραφούν, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλε προκλήσει όσον αφορά τι αλλαγέ του κλίματο και όσον αφορά τους φυσικούς πόρους την ανακύκλωση και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να λαμβάνει η χώρα ο κύκλος της ζωής. Η γεωργία δεν πρέπει να θεωρείται μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα, δεν είναι σωστή προσέγγιση. Όταν μιλάμε για γεωργία, όταν μιλάμε για δασοκομεία, γνωρίζουμε ότι αυτοί οι τομεί είναι ίσως βασικές λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ κυρία Πόλσεν, εξ των Πρασίνων, ο κύριος Χόσλινγκ για δύο λεπτά. Äh Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, αγαπητέ ε, ε, George Lyon, καταρχήν ευχαριστώ για την έκθεση. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά με εσά σαν εισηγητή και βρήκαμε έναν καλό συμβιβασμό τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε και πρέπει το Κοινοβούλιο να μιλήσει με μία ηχηρά φωνή στον τομέα αυτό για να μπορέσουμε να ε, ρυθμίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική. Βεβαίως στους συμβιβασμούς δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε όλα τα θέματα που μας απασχολούσαν αλλά πρέπει να τονίσω ότι χρειαζόμαστε μια πιο πράσινη γεωργική πολιτική και όχι μόνο από πλευράς πολιτικής αλλά και από πλευράς γεωργικής και δεν πρέπει ο ανταγωνισμός να απευθύνεται μόνο ή στην διεθνή αγορά αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα πρέπει να καθορίσουμε τους σωστούς όρους ανταγωνισμού ε, στην Ευρώπη και να μην ε, ε, προσάπτουμε τις ευθύνες της πολιτικής του ΠΟΕ αλλά και εδώ στην Ευρώπη. Επίσης ο πρώτος πυλώνας στο μέλλον θα πρέπει να ρίξει μία σωστή γεωργική πολιτική και να υπάρξει και σωστή κοινωνική πολιτική. Βέβαια αυτό το οποίο δεν θα δεχθούμε είναι ότι η ε, γεωργική μας πολιτική πρέπει να στραφεί προς ε, τις εξαγωγές και θα γινόμαστε όλο και πιο κριτικοί στο σημείο αυτό. Θα θέλαμε να μην υπάρξει η βιομηχανοποίηση της γεωργίας, μια πολιτική γεωργική στραμμένη προς τον ανταγωνισμό, αλλά θα θέλαμε μια πολιτική στραμμένη ε, προς το μέλλον για την ύπεθρο, για την εξασφάλιση των ε, εδαφών του νερού, της ε, βιοπικιλότητος, για την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών και βεβαίως το πιο βασικό σημείο είναι εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ. Εξ των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Τζιμ Νίκολσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να περιγράψει τι απόψει του έναντι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνει προτάσει για το μέλλον τη κοινωνική πολιτική μέχρι το τέλο του έτου να εφαρμοστούν αυτέ οι λύσει. Εγώ και η ομάδα μου θα υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση, αλλά θα ήθελα να πω ότι κάποια τμήματα αυτή δεν μα βρίσκουν συμφώνου και ε, η δομή του δευτέρου πυλώνα θα πρέπει να διατηρηθεί. Είναι κάτι που είναι κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τη ΚΑΠ. Όμω. Εν γέννη πιστεύω ότι είναι μια καλή αφετηρία αυτή η έκθεση για μια συνολική συζήτηση επί του θέματος αυτού, κάτι που δείχνει ότι η Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί. Είχαμε μεγάλη ευθύνη σαν Κοινοβούλιο. Έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι οδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση εξασφαλίζει ότι η γεωργία σαν τομέα μπορεί να είναι ανταγωνιστικό και μπορεί να επιβιώσει στο μέλλον. Η ΚΑΠ είδε τεράστιε αλλαγέ και εμεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στον 21ο αιώνα η ΚΑΠ. Η ΚΑΠ δεν αφορά μόνο τους γεωργούς, είναι και το θέμα ασφαλείας των τροφίμων και την παραγωγή άλλων δημοσίων αγαθών και περιβαλλοντικά ωφέλη και για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους θα πρέπει να διτήσουμε σωστή προσέγγιση. Και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την έξοχη αυτή έκθεση και συνεργασία του. Ευχαριστώ εκ μέρους της Ενωτικής Αριστεράς για ένα λεπτό, κ. Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για το χθεσινό αποτέλεσμα. Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική έχει καταλήξει στην δημιουργία τεράστιων ανισοτήτων, έχουν εξαφανιστεί μέτρα και εργαλεία ε, τα οποία απένιμαν κάποια δικαιοσύνη. Ε, επιβλήθηκαν κάποιοι κανόνες ε, οι οποίοι κατέστρεψαν ε, εκατομμύ... ε, χιλιάδες μικρομεσαίους ε, γεωργούς. Ε. Ξέρουμε λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις από αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρξει μια σε βάθος αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής, μια μεταρρύθμιση της, δίνοντας δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τις Δυνατότητέ τους για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Χρειάζεται να διαφοροποιηθεί η παραγωγή και να υπάρξει μεγαλύτερη διάχυση των προϊόντων και των καλλιεργειών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα εγγυηθούν τις δίκαιες τιμές για την ανταμοιβή ε, των ε, Γιώργων. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος, κύριος Φοντάνα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Λάιον για την εργασία του αλλά και με τον Πρόεδρο και τη της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσόλος ε, διότι συνεργάστηκε άψογα με την Επιτροπή Γεωργίας και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εύχομαι και στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτήν την ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδει στους ε, Γιώργους για να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα αυτό. Ε, η περιοχή από την οποία προέρχομαι, δηλαδή το Βένετο της Ιταλίας, ε, έχει 150 χιλιάδες γεωργικές εκμεταλλεύσεις Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πλούτο που θα πρέπει όχι μόνο να προστατευτεί, αλλά και να του δοθούν περαιτέρω κίνητρα. Αλλά για να μπορέσουν να ασκούν τι λατρεριώτε, οι γεωργοί μα απαιτούν μεγαλύτερη ε, προστασία από την ε, μεταβλητότητα των τιμών. Επίση, σημαντικό είναι να διατηρηθεί και ο δεύτερο πυλώνα τη ΚΑΠ η πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να διατηρηθεί διότι προωθεί τις ε, τοπικές ε, γεωργικές δραστηριότητε, οι οποίες καλούνται να τηρούν κάποια πρότυπα όλο και υψηλότερα. Οι γεωργοί μας ε, ζητούν να υπάρξει μείωση της γραφειοκρατίας την οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά και που συμβάλλει στη μείωση της ανταγωνιστικότητάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φοντάνα και ολοκληρώνουμε αυτόν τον γύρο των αγορητών με την παρέμβαση της κυρίας Ντότζ που εξ ονόματος στο μία εγγραμμένων έχει 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την έκθεση. Ε, ήταν καλό να, που μας άκουγε ε, ο εισηγητή πήγε στα κάτι μέλη για να ακούσει τα προβλήματα και βλέπουμε τα αποτελέσματα τη έκθεση. Το μέλλον τη γεωργία και η ΚΑΠ θα πρέπει να δώσει στου γεωργού ένα ασφαλέ και βιώσιμο εισόδημα. Και οι πληρωμέ του πυλώνα 1 θα πρέπει να ακολουθούν να δίνουν στου αγρότε άμεσε πληρωμέ που θα του δίνει ένα ελάχιστο επίπεδο ασφαλεία εισοδήματο. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ένα προπολογισμό τη ΚΑΠ που θα διατηρηθεί τουλάχιστον στο παρόν επίπεδο και ακόμα πιο σημαντικό να αυξηθεί για να λάβουμε υπόψη την επέκταση της ενώσεως. Η πτυτικότητα των αγορών ήταν εις βάρος των αγορών στην Ευρώπη και θα πρέπει να παραμείνουν τα δίκτυα ασφαλείας, να παραμείνει η σταθερότητα και να εξασφαλιστεί η κερδοφορία. Η διανομή των πόρων για την ΚΑΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κόστος της παραγωγής στα κράτη-μέλη. Ο ορισμός του δικαίου είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί λεπτομερέστερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πληρωμή με βάση την έκταση θα οδηγήσει στο ότι οι αγρότες της ε, ε, Βορείου Ιρλανδίας να παίρνουν λιγότερα χρήματα από την πληρωμή κατά εκμετάλλευση ε, και θα είναι πολύ εις βάρος των γεωργών. Είναι γεωργοί στην Ιρλανδία που έχουν πολύ μικρή έκταση και καλλιεργούν εντατικά και μια τέτοια πληρωμή δεν θα, θα του βοηθήσει να αντιμετωπίσουν το οικονομικό βάρο που έχουν επομιστεί. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γεωγραφική ποικιλομορφία και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην όλη πολιτική θα ακολουθηθεί στην ΚΑΠ μετά το 2013. Και τώρα περνάμε στον επόμενο γύρο των ομιλιών. Πρώτος ο κύριος Δέσσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, <clears throat> κύριε Τσιόλος, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα έχουμε μια σημαντική συζήτηση για την έκθεση Λάιον και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο George Λάιτον για την προθυμία του να συμβιβαστεί σχετικά με την έκθεση αυτή και νομίζω ότι καταφέραμε μεταξύ πολλών πολιτικών ομάδων να έχουμε καλούς συμβιβασμούς οι οποίοι θα επιτύχουν σήμερα το απόγευμα ευρεία συνέχεια συνένεση στην ψηφοφορία. Το θέμα αυτό για την Ευρώπη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της διαδικασίας ενοποίησεως και θεωρούμε στην έκθεση αυτή ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στη Γεωργία μετά το 2013 διότι παράγουμε πολύτιμα τρόφιμα, διατηρούμε ε, ε, θέσεις εργασίας στην βιοτυπική ποικιλότητα, προωθούμε εναλλακτικά καύσιμα αλλά και ε, πρώτες ύλες. Για να μπορούμε όμως να καλύπτουμε και στο μέλλον την πληθώρα των καθηκόντων μας θα πρέπει μετά από το 2013 να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση αυτών των στόχων και γι' αυτό χαιρετίζω την ε, επιθυμία της Επιτροπής να στηρίξει την πολιτική σε δύο πυλώνες. Καταρχήν ε, μία, έναν πρώτο πυλώνα που βασίζεται στη σχέση της γεωργίας με τις άλλες περιοχές και ε, σε ένα δεύτερο πυλώνα ε, για να μπορέσει στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να χρηματοδοτηθεί η πολιτική αυτή και ευχαριστώ εν ονόματι του ΕΛΚ. Ο κύριος Κάπουλα Άντο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, τη συνάδελφη. Οι σοσιαλιστές είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι διότι οι σημαντικότερες προτάσει τους συμπεριλήφθηκαν. 80-90% των τροπολογιών μας ελήφθηκαν υπόψη και Έχουμε προσυπογράψει 49 από τις 50 συμβαστικές προτάσεις στην Επιτροπή Γεωργίας. Φράζουμε την ικανοποίησή μας λοιπόν για το γεγονός ότι η έκθεση ΛΑΙΟΝ δηλώνει ότι επιθυμεί να διατηρηθεί ο κοινωτικός χαρακτήρας της ΚΑΠ και να έχει επαρκή χρηματοδότηση το ζήτημα των ενισχύσεων προς τους γεωργούς αντικαθίσταται με κάποια κριτήρια περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Ε, το να υπάρξει μια πιο ισότιμη και πια δίκαιη κατανομή της, ε, των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων είναι κάτι που μας ικανοποιεί. το η ρύθμιση των αγορών και η διαχείριση των κρίσεων θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να εφαρμοστούν. Νομίζουμε ότι με αυτή την έκθεση περιορίζουμε σημαντικά επίσης και την γραφειοκρατία. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία που μας ικανοποιούν και στα οποία θα πρέπει να στηρίζεται η πρόταση της Κομισιόν που θα υποβληθεί τον Νοέμβριο. Και χαίρομαι επίσης που ο κ. Επίτροπος δήλωσε πρόθυμος να δεχτεί τις συστάσεις μας. Ελπίζω να μπορέσω να συγχαρώ τον Επίτροπο και όλους για του προσεχεί μήνε. Προς το παρόν ευχαριστώ τον συνάδελφο Λάιον, ο οποίο ενισχύει το ρόλο του Κοινοβουλίου ε, τη στιγμή που μέσω της συνθήκης Λισαβόνη αποκτούμε σημαντικότερες εξουσίες. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Ραιμερ, έχει το λόγο. Ξενόματο των Φιλελευθέρων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή συνεργασία και τα βασικά θέματα τα οποία τόνισε η έκθεσή του για το μέλλον της γεωργίας μετά το 2013. Ε, δεν θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τη γεωργία μας, διότι ιδίω ε, πρέπει να καλύψουμε την παραγωγή τροφίμων για τους πολίτες μας, να υπάρχει μία ίση ανάπτυξη για μία διασύνθεση των πόρων ε, με ε, αυτούς οι οποίοι ε, παράγουν. Οι γεωργοί καλούνται να παράγουν περισσότερα με λιγότερους πόρους και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσουν το αναγκαίο πλαίσιο. Αν θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη γεωργία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των γεωργών. Μείωση της ε, ε, γραφειοκρατίας όσο χρειάζεται και καλύτερη αμοιβή για να μπορέσουν να έχουν ικανοποιητικό εισόδημα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λέω ο κύριος Σμίθα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ δεν θα με εξαίρεσα. Συγχαρώ τον Σκοτσέζο συνάδελφό μου τον Τζορτζ Λάιον για μια πολύ καλή έκθεση και μπορούμε να ικανοποιηθούμε πολλά στοιχεία τη εκθέσεω και συμφωνώ με πολλά σχόλια από του συναδέλφου που ακούστηκαν σήμερα. Μου αρέσει ιδιαίτερα η σαφή αναφορά που λέει ότι η πρωταρχικό στόχο τη κοινή ερωτική πολιτική είναι παραγωγή τροφίμων. Όλα τα άλλα είναι αξιόλογα και επιθυμητά, αλλά δευτερευούση σημασία. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό και στο μυαλό μα ότι η επιστημιστική ασφάλεια είναι απόσταση στο τμήμα τη ευρωπαϊκή εθνική ασφαλεία και πρωταρχικό όφελο όφελος της ΚΑΠ και θα πρέπει αυτό να το θεωρήσουμε σαν σκοπό, αυτό σκοπό. Ε, σε αυτό που είπε ο κύριο Λαβία όσον αφορά τον προπολογισμό, κάτι που το υποστήριξαν πολύ λίγοι σήμερα. Σω είναι στερεότυπο σκοτσέζικο να εστιάζεται κανείς το χρήμα, αλλά αν δεν έχουμε επαρκείς νομισματικού πόρου που θετήθεται για την υλοποίηση τη πολιτική αυτή, όλα δεν, έχουν, δεν έχει κανένα νόημα. Και θα ήθελε ο Επίτροπος να μα πει κάποια λόγια πώ θα υπερασπιστεί τον προπολογισμό. Και πολλά κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένη τη Βρετανία θέλουν να σταματήσουν τι άμεσε πληρωμέ προ του γεωργού αλλά θα σα υποστηρίξει το Κοινοβούλιο για σωστό προπολογισμό, σωστή ΚΑΠ και πιστεύω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί σωστή βάση συνεχιζόμενη συζήτηση. Ευχαριστώ και Σμιθ. Για ένα λεπτό το λόγο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου στον ε, κύριο Λάιον διότι εδώ εμφανίζεται το όραμα το οποίο διατυπώνεται για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρέπει να εξισώσουμε ε, το επίπεδο των επιδοτήσεων και αν δούμε ποια είναι η μορφή των επιδοτήσεων βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή ε, υπάρχουν περιοχές που δίδονται 500 ευρώ ανά εκτάριο και περιοχές όπου δίνονται 100 ε, ευρώ ή και λιγότερο ανά εκτάριο. Αυτό λοιπόν πρέπει να εξισωθεί διότι μακροπρόθεσμα δεν πρέπει να διατηρηθούν αυτές οι διαφορές. Ευχαριστώ τον εισηγητή που αντελήφθη αυτό το δημοσιονομικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί χωρίς μία ριζική αναμόρφωση του προϋπολογισμού διότι υπάρχουν ορισμένοι που πρέπει να έχουν κάτι παραπάνω από τους άλλους διότι δεν έχουμε πρόβλημα με την ελευθερία αλλά όπως λένε οι Γάλλοι χρειαζόμαστε περισσότερη αδελφοσύνη για να μπορέσουμε να εξισώσουμε την ελευθερία με την αδελφοσύνη. Η κυρία Ντεμπρούν για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε αυτή την σημαντική έκθεση αλλά απογοητεύτηκα και λίγο διαβάζοντάς τη, διότι δεν καταφέρνει να καθορίσει ένα κάποιο όραμα για την ΚΑΠ που θα, θα οδηγήσει σε αποφυγή της απερίμωσης των εκμεταλλεύσεων και να μπορούν να παράγουν οι γεωργοί τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ζητάει η κοινωνία. Χρειαζόμαστε μια ΚΑΠ που θα εξασφαλίζει ποιοτικά προϊόντα, ποιοτικά τρόφιμα, σε υψηλό επίπεδο, σε υψηλές προδιαγραφές, συντήρηση των εδαφών, προστασία των υδάτων, βιοπικιλομορφία, να εξασφαλίζεται η απασχόληση στην Ήπεθρο και να ενισχύει η οικονομία της Ήπεθρου και να ενισχυθεί επίσης και η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Η ΚΑΠ χρειάζεται μεταρρύθμιση ούτω ώστε να βοηθηθούν εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. για την ώρα το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων πηγαίνει προς τους μεγάλους γεωκτήμονες και τους μεγάλους παραγωγούς. Επίσης χρειαζόμαστε όπως σας είπα τα σωστά κονδύλια για την ΚΑΠ και ευχαριστώ τον κύριο Λάγκη την έκθεσή του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζανκάρλο Σκότα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Λάιον, κύριε Πρόεδρε, εξαιρετικοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Σε ένα πλαίσιο όπως το σημερινό, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν ανάγκη από σημαντική υποστήριξη. Η μορφή του γεωργού απαιτεί σημαντικές εξελίξεις να αναδιαθρώσεις. Ο γεωργός γίνεται επιχειρηματίας ε, στην γεωργία με τις νέες συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να ανακτηθούν και δια, ε, διάφορα εδάφη τα οποία εγκαταλείφθηκαν. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει μια διασύνδεση αυτών των ε, εκμεταλλεύσεων με τις αγορές. Αυτό θα πρέπει να διαδοθεί το σύστημα. Τώρα, στην ορισμό της ΚΑΠ, η Κομισιόν θα πρέπει να υποστηρίξει τη δημιουργία αγροτικών συνεταιρισμών για να καταστούν πλέον ανταγωνιστικοί. Η Κομισιόν θα πρέπει να καθορίσει ένα συγκεκριμένο προπολογισμό για να επιτύχει αυτού του στόχου. Είναι απαραίτητο η χρηματοδότηση τη νέα ΚΑΠ να συνδέονται με τα αποτελέσματα ώστε να αποφύγονται κερδοσκοπίε και σπατάλε. Σε αυτή την περίοδο κρίση, πολλοί νέοι θέλουν να επιστρέψουν στην γη, στη Γεωργία, αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα το ε, υγιές κοστίζουν πάρα πολύ και λοιπά και λοιπά. Επίσης υπάρχει και, υπάρχουν και προβλήματα τα οποία παράλληλα εμποδίζουν τους νέους να ε, επιστρέψουν στις, ε, στον τομέα της γεωργίας. Ως εκ λοιπόν χρειάζεται να προλευθεί κονδύλια για ενίσχυση των νέων. Επίσης χρειάζεται να γίνει και ενημέρωση ξεκινώντα ήδη από τα διακόπτει ο πρόεδρος τον αγορητή. Το λόγο για 1,5 λεπτό έχει ο κύριος Νικουλέσκου. Το Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, να επενέσω την έκθεση για την ποιότητά της και θα ήθελα να υπογραμμίσω και ότι επέφερε συνένεση στην Επιτροπή Γεωργίας. Είναι πολύ φιλόδοξη έκθεση. Προσπαθεί να βρει λύσεις ε, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται. Ταυτόχρονα είναι και ισορροπημένη έκθεση. Προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των νέων κρατών μελών που προσπαθούν να ωφεληθούν από την ΚΑΠ. Επιμένω από τον άρθρο αυτών που αναφέρονται στην αρχιτεκτονική της ΚΑΠ η ΚΑΠ θα πρέπει να βασίζεται επί των δύο πυλώνων που αναφέρονται. Η εξάλληψη αυτών των πυλώνων θα μεταμόρφωνε την ΚΑΠ σε μια πολιτική που δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ανταγωνιστικότητα στη Γεωργία. Η εξάλληψη του πυλώνα για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα καθεστούσε ανέφικτο τα νέα κράτη-μέλη να μπορούν να αναπτύξουν αυτό το νέο κομμάτι της Γεωργίας. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να υπάρχει ένα προπολογισμό που να ταιριάζει, να είναι στα επίπεδα του παρόντο προπολογισμού. Τα νέα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να αυξήσουν την ποιότητα της παραγωγής, κάτι που θα αντικατοπτρίζεται και στην ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε στην Ευρώπη. Για να πετύχουμε αυτά τα επίπεδα θα πρέπει να τύχουν υποστήριξη οι και μια καλά χρηματοδοτούμενη κάψιμενη μένει επιστημιστική ασφάλεια και καλά τρόφιμα για τους Ευρωπαίους. Υπερψηφίζοντας αυτή την έκθεση, το Κοινοβούλιο θα στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη θέση μας που είμαστε εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεκάστρο, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιών Πιστάρδη, τα επόμενα έτη οι προκλήσει που θα ακολουθήσουν τι εξελίξει στον γεωργικό κλάδο θα είναι τεράστιε. Να ικανοποιήσουμε μια αυξανόμενη ανάγκη τροφίμων είναι ε, κάτι το απαραίτητο, θα είναι κάτι το πολύ προβληματικό, διότι θα πρέπει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον παράλληλα. Η Γεωργία λοιπόν αποκτά μια νέα στρατηγική σημασία. Να δημιουργήσουμε την ΚΑΠ του μέλλοντος αποτελεί σήμερα την απάντηση σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις που ε, θα αντιμετωπίσει η κοινωνία μας. Χρειάζεται λοιπόν να απαντήσουμε ήδη στις επιστηστικές ανάγκες του μέλλοντος. Αυτός είναι ο δύσκολος στόχος λοιπόν, τον οποίο θα πρέπει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Γεωργία, το προσεχέται. Μετά από αυτά τα λόγια να πω ότι η Επιτροπή Γεωργίας της οποίας προεδρεύω ε, έκανε μια πολύ εντατική εργασία, ο συνάδελφος George Lyon με την συνεργασία όλων των ομάδων, των πολιτικών ε, μας οδήγησε σε αυτήν εδώ την έκθεση. με έκθεση που είμαστε πεπισμένοι πως θα βοηθήσει στο να διατηρήσουμε τις βάσεις της ε, ΚΑΠ ε, για το, στο μέλλον και θα προετοιμάσει την ανακοίνωση της Κομισιόν για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άιουόρντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου τον George Λάιον για την έξοχη έκθεσή του η ΚΑΠ αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Σε μια μεγάλη Ευρώπη θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει σωστή αγροτική πολιτική με τους αναγκαίους πόρου, ούτω ώστε και στην κοινωνία και στην ύπεθρο και στους αγρότες θα δίνουν τα σωστά αποτελέσματα της ασφαλής στην επιστημική ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να υπάρξει επανεθνικοποίηση της συγχρηματοδοτήσεω θα πρέπει η κοινή αγροτική πολιτική να παραμείνει ευρωπαϊκή πολιτική. Τα τελευταία 50 χρόνια η ΚΑΠ αύξησε την παραγωγικότητα, συνέβαλε σε δικαιότερο επίπεδο διαβίωση για τη γεωργική κοινότητα, εξασφάλισε τη διάθεση των τροφίμων και έδωσε στου καταναλωτέ ποιοτικά τρόφιμα σε λογικέ τιμέ. Οι Ευρωπαίοι πολίτε ωφελήθηκαν σημαντικά από τη γεωργία από τη μορφή τη επιστημική ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντο, καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο, διατήρηση των κοινωνιών τη και υποστήριξη των αγροτικών κοινωνιών. Για να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι η ΚΑΠ και για να αντιμετωπιστούν οι νέε προκλήσει, θα πρέπει να υποστηριχθεί πάρα πολύ, άρα χρειάζεται και μεγάλο υπολογισμό. Δεύτερον, διαφάνεια και αναλογικότητα θα πρέπει να στο επίκεντρο μελλοντική ΚΑΠ. Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική υποστηρίζει του γεωργού. Ο βασικό στόχο είναι να παράγουν τρόφιμα υψηλή ποιότητα και δεν θα πρέπει να του αυξήσουμε διοικητικό άχθο και την γραφειοκρατία. Οι Ευρωπαίοι Γεωργίε για να παράγουν τρόφιμα με την ύψιστη ποιότητα θα πρέπει να παράγουν τον σωστό τρόπο και να υπάρχουν ισότιμε συνθήκε, δίκαιο ανταγωνισμό για τη μελλοντική βιωσιμότητα τη Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Φάιμον για ένα λεπτό έχει οι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη αδικία της τωρινής γεωργικής πολιτικής είναι ότι οι επιδοτήσεις μοιράζονται άνισα μεταξύ των παλαιών και νέων κρατών μελών. Στα νέα κράτη-μέλη εφέτος οι γεωργοί θα πάρουν μόνο 70% από ό,τι παίρνουν οι γεωργοί των παλαιών κρατών κρατών μελών και οι Βούλγαροι μόνο 40% ενώ όλοι εργάζονται στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι αυτή η αδικία θα διορθωθεί άμεσα. Χρειάζονται οι ίδιες συνθήκες ε, για την διανομή των επιδοτήσεων και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το σημείο 6 της εκθέσεως και ελπίζω ότι θα το στηρίξουν και οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κ. Ζαραφιλίδης. Πρόεδρε, η κοινή αγροτική πολιτική σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την αυτονομία της Ευρώπης στην παραγωγή τροφίμων. Στη δεκαετία του 70 σχεδόν το 70% του προπολογισμού της ΕΕ πήγαινε στη γεωργία. Όμως μετά από μια σειρά ανταγωνιστικών μεταρρυθμίσεων οι γεωργικές δαπάνες στον προϋπολογισμό έπεσαν στο 35% για την οικονομική περίοδο 7-13 δυστυχώ σήμερα η αναθεωρημένη καπ σχεδιάζεται με τι ίδιε συνθήκε ανταγωνιστικότητα τη προηγούμενη πολιτική. είναι πρόκληση με το πρόσχημα τη οικονομική κρίση να αποκόβονται οι παροχέ από του αγρότε άλλωστε είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται για τι σημερινέ συνθήκε κρίση. βασικό σκοπό τη νέα καπ θα πρέπει να είναι η προώθηση ενό παραγωγικού μοντέλου συμβατού με την υγιεινή διατροφή την προστασία του περιβάλλοντο και την καταπολέμηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα να μην ξεχνάμε ότι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές σοβαρές ευθύνες έχει το αγροχημικό μοντέλο της συμβατικής γεωργίας το οποίο θα πρέπει να αλλάξει ακριβώς επειδή είναι κατά των αγροτών των λαών και της βιοποικιλότητας του πλανήτη. <clears throat> Εγώ σαν Γεωργός ενδιαφερόμαι το θέμα. Τα σχέδια των μέλλον της ΚΑΠ θα πρέπει να εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο, να λειτουργούν και θα πρέπει να μπορούν να πληρωθούν. Οι στατιωτικοί κάτι λένε. Ε, ε, ε, ότι πρέπει να κάνουν τα σωστά πράγματα. Η ομάδα του ΑΕΛ καταψήφισε την έκθεση στην Επιτροπή, διότι στο σημερινό οικονομικό κλώμα, ε, κλίμα, ενησυχούμε για το κλίμα και οι μη γεωργικοί στόχοι στον πυλώνα 2 παίρνουν πόρους από τους γεωργούς έχει μανία με την αλλαγή του κλίματο η έκθεση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει να δεχθούμε συμβουλέ και να πρέπει τελικά <laughs> αυτοί που καλλιεργούν τη γη να πρέπει να προσπαθούν να στείλουν τι εξατμίσει από τα τρακτέρ κάτω από το έδαφο για να αποφύγουμε την αλλαγή του κλίματο. Και ίσω τελικά θα πρέπει να προσέξουμε και τα ύδατα. Δεν θέλουμε να είναι βρώμικο το νερό. Και οι κτηνοτρόφοι ίσω τελικά θα πρέπει να μειώσουν τι εκπομπέ στο μεθανείο αντικαθιστώντα τελικά τι ζωοτροφέ με πιο ακριβά ε, δημητριακά. Αν πρέπει να υπάρξει ΚΑΠ, θα πρέπει να βοηθά του γεωργού και όχι να του εμποδίζει τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, και κύριοι. Του προσεχεί μήνε θα συζητήσουμε το, τη νέα κοινή πολιτική. Θα πρέπει να πετύχουμε μια καλή συμφωνία και ελπίζω η Βελική Προεδρία να πετύχει αυτό το οποίο δεν πέτυχε η Ισπανική Προεδρία, δηλαδή τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν ε, να διατηρήσουν στο μέλλον μια γεωργική πολιτική η οποία θα είναι πραγματικά ισχυρή με έναν επαρκή προπολογισμό για να αντιμετωπίσουν τι ανάγκε των 27 κρατών μελών, τόσο των νέων όσο και των παλαιών. Και όχι όπω το 2005 όπου έλειψαν τα κονδύλια και χρειάστηκε να βρούμε το θέμα τη διαμόρφωση. Ε, μιλάμε για έναν κλάδο που όχι μόνο προσφέρει ε, προϊόντα, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσει και την, ε, ε, σε τρόφιμα την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προστατεύσει και το περιβάλλον. Χρειάζεται λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μια εγγύηση ασφάλειας επιστηστικής. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος της προσεχούς μεταρρύθμισης, χωρίς όμως να ξεχνάμε την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ η ταχύτητα με την οποία διαβάσατε κυρία Εράνς δυσκόλεψε πάρα πολύ τους διερμηνείς και ορισμένες καμπίνες χρειάστηκε να κλείσουν το μικρόφωνο. Παρακαλώ να προσέχετε πώς διαβάζετε προκειμένου να ακούγεστε και να γίνεστε κατανοητοί. Ο κύριος Λεφόλ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, είχατε μία σύντομη αλλά ευτυχή νύχτα και ε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Επίτροπο αλλά και τον εισηγητή για την έκθεσή του σήμερα το πρωί. Η πρόκληση είναι ότι η γεωργία, η διατροφή και το περιβάλλον αποτελούν αυτή τη στιγμή μία πρόκληση για ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν πρέπει να ε, επανεθνικοποιηθεί η κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει η χρηματοδότηση να είναι στο ύψος των απαιτήσεων και των αναγκών της διατροφικής ε, γεωργίας. Να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει της κοινωνίας και να αποφύγουμε την ε, αστάθεια των αγορών. Και ε, γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε και περαιτέρω. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Θέλω να προειδοποιήσω όλους αυτού που προσπίζουν αυτή τη δομή διότι από ο πλευράς δημοσιονομικής έχει μεγάλο βάρος ο πρώτος πληρώνας αλλά εάν μεταφέρουμε στο δεύτερο πυλώνα ορισμένα στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την επανεθνικοποίηση και τελειώνω με μία τελευταία παρατήρηση. Δημιουργήθηκε η κοινή γεωργική πολιτική στις αρχές της ΕΟΚ και θα πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Λεφόρο. Ο κύριος Άσουρ έχει το λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπε, ο κόσμος αλλάζει και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό η ΚΑΠ να εξακολουθήσει τις αλλαγές, ούτω ώστε να μπορεί να ταιριάζει στις μελλοντικέ προκλήσεις και να μην ζει στο παρελθόν. Η μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ θα έχει ζωτικά σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει αντιμετωπίζοντα θέματα όπω η επιστημική ασφάλεια, η πτυτικότητα των αγορών και η αλλαγή του κλίματο. Θα ήθελα να αναφέρω τρει άλλε αρχέ που κατά την άποψή μου είναι εξίσου σημαντικέ. Πρώτον, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο καλύτερο τρόπο να πετύχουμε του στόχου τη ΚΑΠ είναι να δημιουργήσουμε βιώσιμη δυναμική γεωργία. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε σαν στόχο. Δεύτερον, για να το πετύχουμε αυτό, η ΚΑΠ πρέπει να είναι απλούστερη, δικαιότερη και διαφανέστερη στο τελικό σημείο επιτόπου. Και τέλος κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να δίνει αξία για τα χρήματα που διατίθενται. Όλοι οι τομείς και όλα τα κράτη αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικές τώρα και πρέπει η Επιτροπή να είναι πολύ ρεαλιστική όσον αφορά τι προσδοκίε που έχει από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Κατά την άποψή μου, τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι θα διατίθενται αποτελεσματικά και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Πρόεδρο εισηγητή παρήγαγε μια έξοχη έκθεση, τον συγχαίρω γι' αυτό και με τα χαρά να υποστηρίξω την έκθεση. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριο Μπαυτό, έχει λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής θα εστιάζεται όλο περισσότερο, ε, θα συνδυάζεται με τις πολιτικές εναλλαγή του κλίματος στην Ουαλία. Τα προγράμματα του πλέον 2 θα ε, αντικαταστούν από στόχου που έχουν την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο και την απορρόφηση του άνθρακο. Χρειάζεται αναδάθρωση, καθαρισμό του ύδατο κλπ. Η μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ μετά το 2013 δεν θα πρέπει να θυσιάσει τον πυλώνα 1 για νέου στόχου του πυλώνα 2. Η ενιαία πληρωμή για του γεωργού είναι ζωτική σημασία που βασίζονται στι επιδοτήσει που θα μπορούσαν ξαφνικά να καταργηθούν. Ε, δεν τους άρεσαν οι πληρωμές πέρσι στους ουαλούς καλλιεργούς. Θα πρέπει να έχουν στο μέλλον νέες αναλλακτικές ή αν δεν υιοθετήσουν τα σχήματα προτείνονται θα τιμωρηθούν. Η Ουαλία έχει ιστορία γεωργίας. Πολλές κοινότητες εξαρτώνται από τη γεωργία. Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ που βασίζονται μόνο στην αλλαγή του κλίματος ίσως υπονομεύσουν τις παραδοσιακές περιοχές που ζουν από τη Γεωργία και η Ουαλία είναι μία από αυτέ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Γκαρθία Πέρεθ, που είναι και η τελευταία ομιλήτρια για αυτόν τον γύρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και χρόνια η ΚΑΠ καταβάλει προσπάθειε προσαρμογή και βρισκόμαστε σε μια νέα φάση αυτή τη μόνιμη μεταρρύθμιση. Κύριε Επίτροπε, η, μετα... η πρόταση, η έκθεση, συγγνώμη, Λάιον αναγνωρίζει ότι η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να συμβάλλει στην ε, ε, ανανέωση της ΚΑΠ. Θέλουμε λοιπόν μια ΚΑΠ αποτελεσματική, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, των περιφερειών, αλλά και την διατήρηση του κοινού χαρακτήρα της. Η πτυτικότητα όμως των αγορών, η μεταβλητότητα των τιμών κλπ. μπορούν να έχουν αρνητικέ επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το εισόδημα των γεωργών. Ζητάμε ένα πραγματικό δίκτυο ασφαλείας. Αλλαγέ θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό της ΚΑΠ και θα πρέπει να υπάρξουν τα κατάλληλα κονδύλια, κατάλληλη βρικοδότηση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σε ένα επίπεδο τουλάχιστον με αυτό του παρελθόντος γιατί οι νέες περικοπές θα μπορούσαν να επηρεάσουν αποτελεσματικότητα. Κύριε Επίτροπε, οι γεωργοί θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προσαρμογής. Οι αλλαγές θα πρέπει να συνοδεύονται από μεταβατικές περιόδους ρεαλιστικές. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Λάιον για τις εργασίες του και όλους τους σκιώδεις ηγητές, διότι μα οδήγησαν σε μια έκθεση με την οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε που θα αποτελέσει ένα θετικό μήνυμα για να καλύψουμε τι ανησυχίε και τι αβεβαιότητε των γεωργών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγκαρθία. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα συνάδελφοι. 23 ζήτησαν το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye. Ο κανονισμός αυτό το οποίο προβλέπει είναι 5 να λάβουν το λόγο. Κοιτάξτε, είχαμε προβλέψει εξάλλου 47 λεπτά για την όλη συζήτηση. Έχουμε φτάσει στα 51, έχουμε ξεπεράσει τον προβλεπόμενο χρόνο και δεν έχει ακόμα λάβει το λόγο ούτε ο εισηγητή ούτε και ο επίτροπο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική και αυτό το δείχνει και ο υψηλότατο αριθμό ε, των συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν σε 10 άτομα, τον διπλάσιο από τον προβλεπόμενο από τον κανονισμό. Ο κ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμεί ξεκινήσαμε με την προπόθεση ότι έπρεπε να καθορίσουμε το μέγεθος των επιδοτήσεων και προσπαθούμε να μην δημιουργήσουμε ε, μία διαφοροποίηση μεταξύ παλαιών και νέων κράτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι εμείς πιστεύουμε ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό ε, των ε, επιχειρήσεων και να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις των γεωργών Λοιπόν, για να μπορεί να υπάρξει και διατροφική ασφάλεια. Θα ήθελα τα μέσα αξιολογήσεως της ρυθμίσεως της αγοράς επίσης να ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν και ορισμένες ιδέες για το μέλλον μετά από το 2013 σχετικά με τις ποσοστώσεις του γάλακτος. Διεκόπη. felicitări raportorului felicitări raportorilor umbră și tuturor celor care. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του όλου του κοιόδου και όλου που συμμετείχαν σε αυτό το σημαντικό αυτό πρόγραμμα για το μέλλον τη ΚΑΠ. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινοτική αγορά θα πρέπει να δράσει ενωμένη, ούτω ώστε να εγγυάται την επιστημιστική ασφάλεια, να προωθήσει τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματο να προωθήσει την έρευνα για να χρησιμοποιηθούν καλύτερα δυνατότητες που διαθέτουμε η ΚΑΠ θα πρέπει να δώσει το κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση της παραγωγής μέσω ανάπτυξης παραγωγικότητας ανταγωνιστικότητας και μέσω εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και έτσι να πετύχουμε τη στατηγική ανεξαρτησία όσον αφορά τον εφοδιασμό στους βασικούς τομείς της παραγωγής. Είναι ζωτική σημασία να διατηρηθούν οι δύο πυλώνες της κοινή αγροτικής πολιτικής με σαφή διαφοροποίηση ο πυλώνα 1 θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό ούτω ώστε να εξασφαλίζει δίκαιη, δίκαιρα επίπεδα διαβίωση για όλου του γεωργού. Ο κύριο Μποβέ έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά τον εισηγητή μας Λάιον με τον οποίο συνεργαστήκαμε όλοι αποτελεσματικά για να προοδεύσουμε και να προχωρήσουμε. Να πω μερικά λόγια τα οποία μας οδηγούν σε μια διαπίστωση ότι η Ευρώπη σήμερα εισάγει πρώτες ε, ύλες ε, στον τομέα της γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια φιλόδοξη πολιτική ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των πολιτών μας σε τρόφιμα έχουμε κατά δεύτερο λόγο μια ΠΑΚ, την οποία, μια ΚΑΠ την οποία θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε, διότι είναι άδικη από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πλευρά. Ή διότι οι γεωργοί ε, λαμβάνουν χαμηλότατα εισοδήματα, δεύτερον διότι οι ενισχύσεις δεν ε, δίνονται δίκαια και από οικολογικής σκοπιάς χρειάζεται μια ΚΑΠ η θα φροντίζει τα εδάφη, διακόπτει τον κύριο Μποβέο πρόεδρος και ο Βαντάλεν έχει το λόγο. Πρόεδρε. Να πω ότι με τις εξελίξεις ε, θα υπάρξουν όλο και λιγότερα χρήματα για την κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων η γεωργική, η γεωργική πολιτική. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε τον εφοδιασμό μας σε τρόφιμα. Επίσης, απαιτούμε καλή ποιότητα αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά είναι δημόσια συλλογικά αγαθά ε, για τα οποία δεν ανταμείβονται πάντα οι γεωργοί μας. Κύριε Πρόεδρε, είναι ουσιώδες να ακολουθήσουμε αυτήν την ε, πορεία. Οι ενισχύσεις ε, χρειάζεται να διατηρηθούν, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την εντατικοποίηση για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταμείψουμε αποτελεσματικά τους γεωργούς. Ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταλάβαμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι πολύ ευαίσθητο τομέα, περίπλοκο ζήτημα. Χρειάζεται υποστήριξη της γεωργίας. Ακόμα και μετά τη διεύρυνση χρειάστηκε αυτό. Αυτό όμως οδήγησε σε δυσανάλογες ε, προσεγγίσεις όσον αφορά την κατανομή της οικονομικής ενισχύσεω για του γεωργού. Πρέπει να έχουμε στόχους και δίκαιους και σαφή κριτήρια, δίκαια κριτήρια ούτω ώστε να πετύχουμε ανταγωνιστική αγορά και καλού όρου, διαβίωσης για όλου του γεωργού, Η οικονομική υποστήριξη πρέπει να μοιραστεί σωστά, ισορροπημένα. Έτσι, όλοι να έχουν το ίδιο δικαίωμα επιδοτήσεων, να μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την τροπολογία παριθμών 6 τη εκθέσεω που βοηθά να εισαχθεί η δικαιοσύνη στο μηχανισμό που υποστηρίζει τη γεωργική παραγωγή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει κυρία Βέρτμαν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η πολιτική χρειάζεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντα υπόψη τι περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Για την Αυστρία χρειάζεται ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα επενδύσεων. Αντιμετωπίζουμε μεγάλε προκλήσεις διότι ε, βλέπουμε ότι θα αυξηθεί ο πληθυσμό στα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους και για να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε η Ευρώπη δεν πρέπει μόνο να συνεργάζεται καλύτερα εσωτερικά αλλά και διεθνώς. Ο κύριος Σον Κέλλη το λόγο. Η σημερινή συζήτηση ήταν πολύ ενθαρρυντική από αυτά που ακούστηκαν για τη Γεωργία το ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι νέοι να μπουν στη Γεωργία ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Ζωτική σημασία. Δεν πρέπει να υπάρξει επανεθνικοποίηση τη Γεωργία. Είπε επίτροπο ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι δύο πυλώνε, διότι χωρί τον πρώτο πυλώνα δεν θα υπάρχει ανάγκη για τον πυλώνα 2. Διότι δεν θα είναι επικερδή ε, η Γεωργία και δεν θα παράγονται τα δημόσια αγαθά. Θα πρέπει να δούμε, όπω υπόθηκε, τι είναι δίκαιο. Λαμβάνοντα υπόψη το κόστο και την αγοραστική δύναμη στην Ένωση. Επίσης ο κύριος Λάινεν αναφέρθηκε στην ιστορική βάση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους γεωργούς τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να σταλεί σαφές μήνυμα, να ξέρουν τι πρόκειται να γίνει, ούτως ώστε να μην ακούνε τις εικασίες και να μην είναι θύματα της κερδοσκοπίας και να αγοράζουν και να κινούνται βάσει του ιστορικού μοντέλου. Θα ήθελα σαφές μήνυμα από τον Επίτροπο, το ταχύτερο δυνατό σχετικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ταραμπέλα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο George Lyon για την εξαιρετική έκθεση. Είναι ένα θετικό βήμα προς την ε, αναδιατύπωση της ε, ΚΑΠ. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό από οικολογικής, περιβαλλοντικής κλπ. Ε, ε, είναι κάτι το οποίο το προσδοκά και ο φορολογούμενος ε, και να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατανομή ανάμεσα στου 27 κράτη και να υπάρχει μια καλύτερη χρησιμοποίηση των δημοσίων πόρων. Ε, ναι, προτάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν για να διασφαλίσουμε την ε, επιστημική ασφάλεια των εργαζομένων. Έχουμε ανάγκη από μια ΚΑΠ η οποία όμως ε, απαιτεί την ικανή χρηματοδότησή της. Ε, τονίζονται οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΚΑΠ, ανεδιαχείριση των υδάτων, βιοπικιλότητα, διάβρωση των υδάτων κλπ. Αυτή η έκθεση θέλει μια ΚΑΠ πιο αποτελεσματική που θα αποκρίνει τις ανάγκες των γεωργών. Κλείνει το μικρόφωνο του ο σας ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Ο κύριος Σιλβέστρης, τον οποίο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την υποδοχή στην υπέροχη περιοχή την οποία επισκεφτήκαμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε η ε, ΚΑΠ θα είναι απαραίτητη και για το μέλλον και για λόγους απασχόλησης. Ξέρουμε ότι στην Ευρώπη ε, η απασχόληση των γεωργίων μειώθηκε κατά 25% και χάθηκαν 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αν θέλουμε λύσεις για την αυξανόμενη και καλπάζουσα ανεργία ε, σταματήσει, θα πρέπει να εγγυηθούμε στην ΚΑΠ ικανούς πόρους για να οδηγηθούμε σε μια ικανοποιητική βελτίωση και ανάπτυξή της. Θα πρέπει να εγγυηθούμε τουλάχιστον το ίδιο αριθμό, ε, τον ίδιο ποσό μάλλον κορδιλίων που είχαμε και στο παρελθόν. Το ζήτημα δεν είναι να, ε, να υπάρξουν πόροι, πρέπει να μην μειωθούν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να χρειάζεται να υπάρξει μια θετική αντιμετώπιση. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν το ε, εισόδημα των γεωργών ε, Διακόπτει τον ομιλητή ο πρόεδρος, ο κ. Άλβης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψηφιζόμαστε μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική που απευθύνεται όχι μόνο προ του γεωργού, αλλά και στου πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε που θέλουμε φιλόδοξο προπολογισμό για να τοποκριθούμε στι προκλήσει ε, και οι προσπάθειες που καταβάλλονται στις περιοχές της Ευρώπης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη γεωργία στην Σαζόρες, που είναι πολύ σημαντική γεωργία για την διαβίωση εκεί πέρα. Θα θα πρέπει να υπάρξουν ιστορικά κριτήρια για τη διανομή των πόρων. Μάλλον, ιστορική βάση για τη διανομή των πόρων ήταν επιβλαβή στου Πορτογάλου καλλιεργητέ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα τη γεωργία, να ρυθμιστεί καλύτερη αγορά και διαχείριση των κινδύνων, να εξασφαλίσουμε μια σωστή λειτουργία τη αγορά και σταθερότητα τη γεωργική παραγωγή. Η κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2013 θα πρέπει να αυξήσει την αναγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, εξασφαλίζοντας την διανομή των προϊόντων στην, στην επισητιστική αλυσίδα. Και του κόβει το το μικρόφωνο. Κοιτάξτε, με ακούτε, με ακούτε, 30 έχουν ζητήσει το λόγο. Και δύο αιτήσει για διαδικαστικό. κυρία Μαγκίνε, διαδικαστικό. Ένα διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε και φαντάζομαι ότι πολλοί συμφωνούν ε, με την διαδικασία Catch the Eye αλλά τα μέλη της Επιτροπής που έχουν δουλέψει καιρό επί του θέματος αυτού νομίζω ότι αξίζουν ε, να διατυπώσουν την άποψή τους. Δεν, ε, έπιασα το... δεν με έπιασε το μάτι σας διότι δεν με κοιτούσατε. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στις λιγότερες προνομιούχους περιοχές οι οποίες ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη και ελπίζω να με στηρίξετε στο θέμα αυτό. Κυρία Μαγκίνες, σχεδόν κατά όλες τις συνεδρίασεις σας κοίταζα. Ε, είδα, ζητήσατε το λόγο όπως και άλλοι συνάδελφοι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο προκειμένου να δώσουμε προτεραιότητα στους συναδέλφους που είναι μέλη της αρμόδιας επιτροπής, αλλά θα δίνω το λόγο σε αυτούς οι οποίοι πρώτοι ε, ζητούν το λόγο και τους πρώτους τους αντιλαμβάνομαι. Ε, ναι, καταρχήν προβλέπονται πέντε σύμφωνα με τον κανονισμό συνάδελφοι να λάβουν το λόγο. Έδωσα το λόγο σε δέκα και φρόντισα να γίνει μια κατανομή ανά πολιτική ομάδα. Να τηρήσω λοιπόν αυτήν την αρχή. Δεν μπορούμε όμως να δώσουμε το λόγο σε όλους όσοι τον ζήτησαν διότι έχουμε συγκεκριμένο χρονικό όριο. Ο κύριος Σόγκορπ το λόγο για διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποθέτω ότι εμένα εννοείται και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η προλαλή σας. Καταρχήν ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη γενναιοδορία σας. Αντιλαμβάνουμε την άποψή σας. Καταλάβετε όμως ότι και εμείς αντιπροσωπεύουμε περιοχές Ευρώπης που είναι πολύ βεβαρημένε Και δεύτερον αναφέρατε ότι το πρόβλημα δεν έχει ρυθεί με τη διαδικασία Catch the Eye. Οπότε θα πρέπει να ρυθμιστεί. Δηλαδή τι γίνεται. Πρέπει να ζητούμε το λόγο μία μέρα πριν ή θα πρέπει να ξεκινήσουμε τρεις μέρες πριν για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Διότι ε, θα έπρεπε να ξέρουμε ποιοι είναι οι δέκα όταν ε, έχουν επιλεγεί και έτσι και εσείς θα είσαστε ε, πιο δίκαιος αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη διαδικασία και θα είσαστε πιο δίκαιος απέναντί μας. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα του catch the eye είναι όπως καταλαβαίνετε υποκειμενικό διότι ο πρόεδρος ε, έχει μάτια αλλά δεν είναι αετήσια τα μάτια αυτά και μερικές φορές ε, στο μάτι του μπαίνουν κάποια άτομα <laughs> κάποια άτομα παρατηρεί, κάποια άτομα βλέπει εντάξει έχετε δίκιο είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί με τρόπο ορθολογικό θα έλεγα από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Παράδειγμα, αυτό που είπε η κυρία Μαγκίνες ότι δηλαδή οι συνάδελφοι της ε, αρμόδιας επιτροπής θα έπρεπε να είχαν προτεραιότητα, εντάξει, κατά την μου έχει δίκιο. Αλλά δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Το μοναδικό που προβλέπεται είναι ο πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος διευθύνει τη συζήτηση και ανάλογα με την εκτίμησή του και με την ανάλογα με τους συναδέλφους φυσικά που τον ζητούν. Δεν, πρόκειται να δώσω σε άλλον τον λόγο. Αλλά οι ε, συνάδελφοι θα πρέπει να ξέρουν ότι το, αυτό το καρτελάκι το θάλασσι δεν ε, χρησιμοποιείται για να παίρνετε το λόγο στην διαδικασία Catch the Eye. Προβλέπετε μόνο για να διακοπεί ε, ένας αγορητής την ώρα που μιλάει και να του γίνει μια ερώτηση διάρκεια 30 δευτερολέπτων. Αλλά εδώ είναι συνάδελφοι οι οποίοι συνεχώ σηκώνουν αυτό το θαλασσί καρτελάκι. Λοιπόν, θα οργανώσουμε λοιπόν ένα σεμινάριο προκειμένου οι συνάδελφοι να καταλάβουν ότι αυτό το θαλασσί χαρτάκι έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αν θέλετε λοιπόν να ε, ζητήσετε το λόγο στο πλαίσιο διαδικασία κάτω διάρκεια, θα σηκώσετε το χέρι σα Δεν θέλω να παρατείνω περαιτέρω τη συζήτηση. Έχουμε λοιπόν σε, όλα, σε όλο αυτό το διάστημα που μιλάω και μιλάτε θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει το λόγο σε άλλα τρία-τέσσερα άτομα. Εμπεστώσει το λόγο και ο κύριος Σιόλος για να απαντήσει. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω εάν υπήρξαν πολλές ερωτήσεις οι οποίες ε, τέθηκαν. Εγώ διεπίστωσα ότι υπήρξαν ιδίως δηλώσεις. Δηλώσεις για ορισμένες αρχές οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην έκθεση. Αυτό που όμως σημείωσα από αυτή την έκθεση είναι ότι χρειαζόμαστε μια κοινή γεωργική πολιτική, μια πολιτική που πρέπει να είναι κοινοτική και χρειαζόμαστε και έναν προπολογισμό ο οποίος να είναι ανάλογος με τους στόχους αυτής της γεωργίας, δηλαδή ένα ρεαλιστικό προπολογισμό, ο οποίος κατά τη γνώμη μου θα ανταποκρίνεται στους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ζητάμε όλο και περισσότερα πράγματα από τους γεωργούς και ζητούμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε να χρησιμοποιούνται καλύτερα και πιο, με μεγαλύτερη διαφάνεια. Ο κύριος Λεβαντόσκι, επίτροπος ε, του προϋπολογισμού είναι εδώ ίσως για να μας επιβεβαιώσει ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα συνάδει με τους στόχους που έχει θέσει. Επίσης, για να μπορέσει η κοινή γεωργική πολιτική να επιτύχει τους στόχους της θα πρέπει να λάβει υπόψη τις διάφορες, τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τομέων της γεωργίας στην Ευρώπη και ιδίως στις περιφέρειες όπου αναπτύσσονται για να επιτύχουμε τους στόχους οι οποίοι να αποβλέπει ε, όχι μόνο στην τροφοδότηση των αγορών αλλά και μία εξέλιξη για μία καλύτερη συνειδητοποίηση ε, του περιβάλλοντος της διαχειρήσεως των φυσικών πόρων των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης στην Ήπεθρο και τον τρόπο με τον οποίο η γεωργία και ε, η διατροφική ε, βιομηχανία μπορεί να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ε, θέλουμε επίσης να συμβάλλουμε στο να ενθαρρύνουμε τους νέους, να τους δώσουμε μία προοπτική για να μπορέσουν να εγκατασταθούν, να επενδύσουν στη γεωργία κατά τρόπον ώστε η γεωργική δραστηριότητα να έχει μέλλον και να επιτύχουμε το στόχο μας. Θα δώσω επίσης και ένα σαφές σήμα και να απαντήσω στον κύριο Κέλλη για τις άμεσες ενισχύσεις διότι για να υπάρχει μια πιο σωστή και δίκαια γεωργία, πιο διάφανη και πιο αποτελεσματική, θα πρέπει να διατυπώσουμε σαφή κριτήρια για την κατανομή αυτών των πόρων και οι ιστορικές αναφορές κατά τη γνώμη μου δεν είναι διάφανο και δίκαιο κριτήριο. Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτές τις ιστορικές αναφορές σε πιο σαφή, με πιο σαφείς στόχους, πράγμα το οποίο θα λάβει υπόψη περισσότερο την ποικιλομορφία της γεωργίας που έχουμε στα κράτη-μέλη και θα επιτρέψει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που διαθέτουμε θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική για την Ευρώπη, για όλη την Ευρώπη, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως μια κοινή γεωργική πολιτική που δεν θα εμποδίσει άλλες περιοχές του κόσμου να αναπτύξουν τη δική τους ε, γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσόλος, λέει ο Πρόεδρος και θα ολοκληρώσουμε την ε, συζήτηση με την παρέμβαση του εισηγητή κ. Λάιον, τον οποίο και συγχαίρω για την εξαιρετική εργασία του. Κύριε Λάιον, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχάς να αναφερθώ σε κάποια από τα βασικά θέματα που έθιξαν οι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Νέα στατηγική σημασία για την παραγωγή των τροφίμων στην ΚΑΠ. Βεβαίως, βεβαίως. Δύο πυλώνες. Ναι, βεβαίως. Συμφωνώ με αυτά παραγωγή τροφίμων στο επίκεντρο της ΚΑΠ. Ναι, και αυτό, περί αυτού πρόκειται η ΚΑΠ. Τα υπόλοιπα είναι προστιθέμενα που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να έχουμε κερδοφόρο αγροτικό τομέα για να μπορέσουμε να έχουμε ωφέλη για το περιβάλλον, να αντιμετωπίσουμε αλλαγή του κλίματο και όλα τα άλλα που αναφέρουμε στην έκθεση. Ισχυρό προπολογισμό. Ναι, βεβαίω. Δίκαιο προ και τα παλιά και τα νέα Πολλά μέλη αναφέρθηκαν σε αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το καλύψουμε και θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και διαφανεί όσον αφορά τη ανομή των πόρων μεταξύ κρατών μελών. Και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσει στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Ένωση του 2020. Θα πρέπει η γεωργία και η κοινή αγροτική πολιτική να ειδωθούν σε ένα κομμάτι τη λύσεως για την επίτευξη αυτών των στόχων και όχι σαν ένα κομμάτι του προβλήματο. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στον Ισελ Ντάντον, τον κύριο Χόσλινγκ, τον κύριο Λέσνιτσακ και τον Τζιμ Νίκολσον, τους ηγητές μου πάρα πολύ καλή συνεργασία που οδήγησε σε ισχυρότατη έκθεση πιστεύω που καθορίζει ένα σαφές όραμα σχετικά με την πορεία που επιθυμεί να ακολουθήσει η ΚΑΠ ε, το Κοινοβούλιο μετά το 2013 και το Κοινοβούλιο βρίσκεται σε ισχυρότατη θέση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο Γεωργίας. Και Επίτροπε βοηθήστε μας και σίγουρα θα πετύχουμε την υλοποίηση αυτού του οράματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάιον. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτηση και όσον αφορά αυτό το θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό και σημαντική η ψηφορία θα γίνει στις 12 και ζητώ συγγνώμη τους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να μιλήσουν.